Επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα έγγραφα τα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Έχετε αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε λάβει μια αίτηση του ΕΛΚ